να αποτίσουμε φόρο σα στα θύματα της σφαγής στην Νορβηγία. Τον Ιούλιο συνέβη αυτό το θλιβερό γεγονός. Επιτρέψτε μου καταρχήν να απευθύνω τις εξής παρατηρήσεις προς εμάς. Πρώτα, θα ήθελα να δώσω μια σύντομη ε, δήλωση. Αν θέλετε μπορείτε να παραμείνετε στα έδρανά σας καθισμένοι, να καθίσετε. Ευχαριστώ. Koleżanki Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κάνουμε λόγο για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας έπληξε και μας συγκλώνησε όλους μας. 22 Ιουλίου η Ευρώπη αποτέλεσε, έγινε θύμα τρομοκρατικής απόπειρας. Στην Νορβηγία ένας εγκληματίας σκότωσε 79 ανθρώπους τα χειρότερα πράγματα συνέβησαν όσον αφορά αυτό το πλήγμα της ε, ξενοφοβίας. Ε, αυτές οι δύο απόπειρε στην Οτόγια και στο Όσλο έπληξαν ε, την Ευρώπη, τους νέους που ονειρευόντουσαν να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Και αυτές οι εγκληματικές πράξεις θα πρέπει με κάθε τρόπο να καταδικαστούν από όλους μας ομόθυμα η μέρα εκείνη κατέδειξε ότι η τρομοκρατία δεν είναι μόνο ένας κίνδυνος εκ των έξω όσον αφορά την Ευρώπη, όπως συνέβη κατά την 11η Σεπτεμβρίου το 2001 στις ΙΠΑ ε, ένα μέλος της ίδιας της κοινωνίας αυτού του κράτους ένας φανατικός με αυτόν τον κτηνόδιωμό τρόπο έπληξε την κοινωνία της Νορβηγίας γι' αυτό πρέπει να συναγάγουμε τα αναγκαία συμπεράσματα από τέτοιου είδους πράξεις αφενός πρέπει να πράξουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε η εσωτερική ολοκλήρωση να επιτευχθεί ώστε όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη και παντού όσοι ζουν σε αυτή την οικουμένη παγκόσμια να μπορέσουν να εκφράσουν εκφράσουν την ικανοποίησή τους και την ευτυχία τους διότι είναι δυνατόν να συμβιώνουμε όλοι από κοινού και να συνεπάρχουμε και πρέπει να συνεργαστούμε με όλες τις χώρες που καταπολεμούν την τρομοκρατία. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή σε μια εποχή της παγκοσμιοποίησης και στην εποχή του διαδικτύου που δεν υπάρχουν σύνορα. Στην Νορβηγία όπου απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης με αυτόν τον τρόπο υπέστη επίθεση η κοινωνία της Νορβηγίας από έναν τρομοκράτη τρομοκρατία όμως ποτέ δεν θα μπορέσει να κλονίσει το σύστημα αρχών και αξιών μας στην Ευρώπη. Ποτέ δεν θα καταφέρει να το υπονομεύσει η ανεκτικότητα, η αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη θα εξακολουθεί να είναι στόχος όλων μας. Εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μας με τον λαό της Νορβηγίας και με την κοινωνία της Νορβηγίας στο σύνολό της. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας στα θύματα και στις οικογένειές τους και οικείους τους. Με αυτές τις σκέψεις εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και ε, συμμετέχουμε στο πένθο σας. Ακόμα και δύο μήνες μετά από αυτή την ε, τραγική πράξη, αυτή την τραγωδία, δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με αυτά. Ευχαριστώ. Και τώρα για παρατηρήσεις ε, των ηγετών των επικεφαλής των ε, κοινοβουλευτικών ομάδων ένα λεπτό φόρου τιμής θα αποτύσσουμε στα θύματα. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τον εκπρόσωπο του ΕΛΚΑ. Εσείς παρακαλώ. Herr Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ θερμά για το ότι μα δίνετε την δυνατότητα εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απευθυνθούμε προ τον λαό τη Νορβηγία και να εκφράσουμε τη θλίψη μα με αυτέ τι παρατηρήσει. Θεωρούμε ότι ο Νορβηγικό λαό είναι ένα αδερφό λαό. Αυτά τα οποία συνέβησαν στην Νορβηγία είναι μια φρικαλαιότητα και δείχνει ότι το κακό, τα δεινά δεν έχουν σύνορα. Οι νέοι, οι νέοι αυτοί που έπεσαν θύματα αυτής της εγκληματικής πράξης που δεν τους γνωρίζουμε. Δεν τους γνωρίζουμε ωστόσο ξέρουμε ποιες, είναι, ποιες ήταν οι ελπίδες τους και η γνώση τους για το καλό και το κακό και η επιθυμία τους να ζουν σε ένα καλύτερο κόσμο. Όλοι μας ε, ε, συγκλονιστήκαμε από αυτά. Ο Χένρικ Ήψεν, ο θεατρικός συγγραφέας της Νορβηγίας, έγραψε, είπε κάποτε τα εξής. Και μάλιστα όταν η Δανία υπέστη τον πόλεμο Σλέσβιχ Χόλσταϊν σε σχέση με την Γερμανία. Είπε θα πρέπει όταν κάποιος κινδυνεύει όλοι να τρέξουν, να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν. Εμείς στην Σουηδία κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτά τα οποία συνέβησαν στην Νορβηγία, στο Όσλο και στην Ούτοια θα πρέπει να δείξουν ότι η υπόθεση αυτή της Νορβηγίας είναι υπόθεση όλων μας. Μας αφορά όλους. Η αλληλεγγύη, η δική μας συμμετοχή σε αυτή τη θλίψη δεν μπορεί να αντισταθμίσει ποτέ βέβαια το πένθος εκείνων που έχασαν τους οικείους τους στην ίδια την Νορβηγία. Όμως ένα πράγμα μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα. Συμμετέχουμε σε αυτό το πένθος σας, στον πόνο σας και η δική σας υπόθεση η δική σας ε, ζωή είναι και δική μας υπόθεση και δική μας ζωή. Ε, από πλευράς ε, Νορβηγού συγγραφέα και που σε πάρα πολλές ε, πένθυμες τέτοιες εκδηλώσεις και κηδείες αναφέρθηκε στην Νορβηγία αυτό το καλοκαίρι θα πρέπει σε σχέση με αυτούς τους νέους και σε σχέση με τα όσα συνέβησαν να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το πένθος. Γράφει για τους νέους. Ο πόλεμος είναι η ίδια η περιφρόνηση της ζωής και γι' αυτό θα πρέπει την δύναμη για την ειρήνη, να χρησιμοποιήσουμε την δύναμή μας υπέρ της ειρήνης. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος τρόπος να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε σχέση με τον νορβηγικό λαό από το να συνεισφέρουμε υπέρ της ειρήνης. Και για το μεγαλόπνο αυτό πνεύμα υπέρ της κοινωνίας κατά του μίσους και κατά του διχασμού. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να μπορέσουμε να πούμε όλοι μας ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί έξω και όλοι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να μας πλήξουν ως τρομοκράτες οι οργανωμένοι ε, στο οργανωμένο έγκλημα δεν μπορούν να μας πλήξουν. Είναι αυτή η δύναμή μας και θα μπορέσουμε να τους πούμε με αυτόν τον τρόπο χάσατε εσείς αυτό το παιχνίδι. Εμείς κερδίζουμε. Θα συνεχίσετε να είσαστε εσείς οι χαμένοι και εμείς θα είμαστε πάντα οι κερδισμένοι γιατί είμαστε υπέρ της ειρήνης και της ομόνοιας. Έτσι μπορούμε να εκφράσουμε με τον καλύτερο τρόπο την αλληλεγγύη μας υπέρ των Νορβηγών και υπέρ των θυμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχετε τον λόγο κύριε Σούλτς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πολλοί από τους φίλους μας στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα πολλές γυναίκες, πολλοί άνδρες από το Διεθνές Σοσιαλιστικό Σοσιαλδημοκρατικό Κίνημα γνωρίζουν αυτό το μέρος πολύ καλά. Δεν είναι η Οτόια μόνο ένα μέρος όπου οι Νορβηγοί Σοσιαλδημοκράτες και όπου οι ε, νέοι σοσιαλιστές συχνά συναντώνται εκεί και περνάνε τις διακοπές μαζί τους. Για πολλούς από τους φίλους μας αυτός ο τόπος συνδέεται με προσωπικά τους βιώματα, με αυτά που έχουν ζήσει προσωπικά εκεί. Ήταν ένα πλήγμα κατά των νέων των σοσιαλδημοκρατών της σοσιαλδημοκρατίας στην Νορβηγία. Όμως ο προλαλής σας το εξέφρασε με καλύτερα λόγια. Ε, ήτανε, είμαστε εμεί τα θύματα, τα θύματα οι νέοι των νέων σοσιαλιστών. Ήταν θύματα ενός δολοφόνου που είχε ως στόχο τους σοσιαλδημοκράτες σε αυτή την περίπτωση. Ήθελε να εξοντώσει αυτός ο ένα ολόκληρο σύστημα αρχών και αξιών. Αυτό ήταν ο στόχο του. Η φρικαλαιότητα αυτού του εγκλήματο έγκυται στο ότι δεν ήθελε αυτό το σύστημα αξιών και αρχών να έχει μέλλον και να επιβιώσει. Και γι' αυτό ιδιαίτερα του νέου αυτού ήθελε να σκοτώσει, να του δολοφονήσει. Συμβολική πράξη να σκοτώσει αυτού του νέου, ώστε αυτή η ιδέα του να μην μπορέσει να ε, συνεχιστεί στο μέλλον, να μην ευδοκιμήσει. Η επίθεση ήταν εις βάρος μιας ιδέας λοιπόν, η ιδέα ήταν ο στόχος. Και αν διαβάσει κανείς τις θέσεις, τα επιχειρήματα αυτού του ατόμου, διαπιστώνει αμέσως ταχύτατα κανείς ότι καμιά ανοιχτή κοινωνία, δεν σέβεται την ανοιχτή κοινωνία, τους άλλους πολιτισμούς, ε, θεωρεί ότι η λευκή είναι ανώτερη από άλλες φυλές, δεν είναι υπέρ της ισότητας των φυλών ε, και της ισότητας άσχετα από το σε ποια φυλή ανήκει κανείς, σε ποια Φιλή και σε ποιο φίλο είναι επίθεση εις βάρος των αρχών και αξιών μας, επίθεση εις βάρος των αξιών όλων μας. Δεν είναι επίθεση μόνο εις βάρος των αξιών των σοσιαλδημοκρατών, είναι εις επίθεση εις βάρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας και των αρχών της. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, μέλη της Ευρωβουλής, εμείς είμαστε εκείνοι που εκπροσωπούμε ως Κοινοβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο, αυτές τις αρχές και αξίες. Ήταν λοιπόν επίθεση εις βάρος μας, εναντίον μας, επίθεση εις βάρος εναντίον όλων μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο να αποτίσει φοροτιμή στα θύματα, αλλά το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο να σκεφτεί ότι οι ίδιες οι δικές μας αρχές και αξίες υφίστανται επίθεση εκ των ένδων από ε, το εσωτερικό της ε, ίδιας της Ένωσης. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να πούμε ότι σε τέτοια επιχειρήματα δεν υπάρχει θέση. Δεν υπάρχει θέση για την μη ανεκτικότητα, για την ε, μυσαλλοδοξία, για την ξενοφοβία, για τον ρατσισμό, για την δίωξη των μειονοτήτων. Δεν μπορούμε να ασκούμε μια πολιτική των <clears throat> αποδιοπομπαίων τράγων αν από κοινού δράσουμε και αντιμετωπίσουμε αυτή την πράξη και αυτούς τους στόχους, τότε θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το κύμα. Αυτό βέβαια δεν είναι καμιά παρηγοριά για τους γονείς, για τα αδέρφια, για τους οικείους εκείνων που έχασαν τους δικούς τους και που υποφέρουν βάθια. Και γι' αυτό εκφράζω και εγώ την ευγνωμοσύνη μου για τα συλληπιτήρια που εκφράσατε εσείς κύριε Πρόεδρε για αυτούς. Πολλές επιστολές έλαβα σε σχέση με αυτή την επίθεση, σε σχέση με τη σοσιαλδημοκρατία και για την Νορβηγία και για τη Διεθνή Σοσιαλδημοκρατία. Πολλέ επιστολέ προήλθαν από αυτό το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Μία θα ήθελα να αναφέρω που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ένα συνάδελφο την συνέταξε και έγραψε και είπε ότι αυτή την επίθεση εις βάρος αυτών των ε, κοριτσιών και των ε, αγοριών είναι μια επίθεση που θεωρεί ότι είναι επίθεση εις βάρος του προσωπικά. Ο κύριος ε, Μάριο Μάουρο το ανέφερε. Το αναφέρω αυτό προσωπικά επειδή δεν είναι σοσιαλδημοκράτης. Είναι αδιάφορο αν είναι κανείς σοσιαλδημοκράτης ε, ή χριστιανοδημοκράτης, αν είναι πιστός χριστιανός ή όχι, αν είναι κανείς λευκός ή όχι, αν είμαι λευκός ή έγχρωμος αν είμαι αριστερός ή δεξιός ε, όταν εργάζομαι ως δημοκράτης. Τέτοιοι τρομοκράτες θέλουν όλους μας να μας εξοντώσουν, να μας εξαφανίσουν και γι' αυτό προς όφελος των Ευρωπαϊκ... της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την οποία συνεργαστήκαμε ως πολυεθνικό, ως πολυθρησκευτικό, ως πολυφιλετικό και πολυπολιτισμικό κοινοβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο, αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτού του είδους τρομοκρατικές πράξεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκίφερ Χόφστατ θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, το 1940 στην αρχή της κατοχής ε, των Ναζί ο Νόραλ Κρίχ, ο νορβηγός ποιητής, είχε πει «Είμαστε πολύ λίγοι σε αυτή τη χώρα και ο καθένας είναι ε, ο καθένας και ακόμη και οι εχθροί είναι αδελφοί φίλοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ζούμε την εποχή που 76 νέοι ε, σφαγιάστηκαν, σκοτώθηκαν νέοι, οι οποίοι συνειδητοποίησαν τι σημαίνει δημοκρατία και το να είσαι πολίτης. Και μερικοί δεν, ήταν, δεν είχαν φτάσει στην ηλικία να ψηφίσουν, ήταν ενήλικοι. Ήταν ένα μεγάλο δράμα, αλλά και κατάφορη επίθεση στη δημοκρατία. Νομίζω όμως ότι το να εκφράζουμε την απέχθειά μας δεν αρκεί. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε μπροστά σε μια βίαιη πράξη όπως εκείνη που έγινε. Ίσως ήταν ένας παράφρον, ίσως ενεργούσε μόνος του, αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Αυτός είναι προϊόν μιας κοινωνίας, ενός κινήματος, μιας κοινότητας, ακτιβιστών, blogger, οι οποίοι απορρίπτουν και απεχθάνονται την κοινωνία μας. Εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο είναι πώς δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί να αποποιούνται κάθε ευθύνη, ενώ θα έπρεπε πρώτοι να αντιδράσουν κατά της ιδεολογίας που βρισκόταν πίσω από την πράξη αυτή. Μια ιδεολογία που είναι αντισλαμιστική, κατά της μετανάστευσης, κατά μιας πολυπολιτισμικής και ποικίλη κοινωνίας, κατά της Ευρώπης και τέλος κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός ο άνθρωπος πράγματι ενεργούσε με βάση μια ιστορία που ακούμε όλο και περισσότερο, που περιγράφει τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη ως δραματική και θεωρεί ότι η κοινωνία μας έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον να ε, ε, έχει κανείς εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε δημοκρατική κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν να επαναλάβουμε τις λέξεις του πρώην Πρόεδρου Κλίντον, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις όταν μίλησε στη 15η επέτειο του βομβαρδισμού στο Κλαχώμας. Είπε ότι εμείς οι πολιτικοί και οι πολιτικοί σχολιαστές είμαστε επίσης υπεύθυνοι για αυτό το γεγονός, επειδή οι λέξεις μας, τα λόγια μας δεν είναι ουδέτερα. Είναι λόγια τα οποία μεταφέρονται στο διάστημα σε όλη την Ιφίλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα ο κύριος Κολμπέντιτ παρακολουθεί. Όταν υπάρχει μια πραγματική σφαγή, οι περισσότεροι από εμά ε, παραμένουν άφωνοι. θυμόμαστε, φοβόμαστε και με την πάροδο του χρόνου αρχίζουμε να σκεπτόμαστε. Γεγονός είναι ότι αυτή η επίθεση που έγινε στην Ορβηγία ήταν εστιασμένη σε νέους, ε, νέοι ε, και δημοκράτες οι οποίοι υποστήριζαν μια ιδέα της αλληλεγγύης ε, πολυπολιτισμικής νέοι οι οποίοι βρισκόταν γύρω από αυτή την ιδέα, είχαν συγκεντρωθεί γύρω από αυτή την ιδέα. Υπήρχαν νέοι Νορβηγοί, κουρδικής καταγωγής, αλλά από κάθε άλλη καταγωγή που έκφραζαν την πολυπολιτισμική κοινωνία, αυτές τις κοινωνίες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και πολιτικοί, εδώ και λίγο καιρό μας λένε, ότι η πολυπολιτισμική κοινωνία έχει χρεοκοπήσει. Και ρωτούσα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εκείνους οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί Νορβηγοί, πραγματικοί Φιλανδοί, θα εκδιωχθούν, πραγματικοί Ολλανδοί, πραγματικοί Γάλλοι, πραγματικοί Σουηδοί, πραγματικοί Ιταλοί, πραγματικοί οτιδήποτε, όλοι αυτοί θα σταλούν πού, πού θα τους στείλετε. Και σε αυτά τα λόγια εξελίσσεται το μίσος αυτό. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι η πραγματικότητα είναι κάτι που μας αγγίζει, που την ασπαζόμαστε όταν μιλάμε ότι πρέπει να προασπίσουμε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τις ευρωπαϊκές αξίες, να προασπίσουμε ε, τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό σημαίνει σε καλά γαλλικά να προασπίσουμε την πολυπολιτισμική ταυτότητα της σημερινής Ευρώπης επειδή αυτή είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα και κατά της ιδέας αυτής έγινε αυτή η σφαγή. Και όταν Έλληνας, ε, με συγχωρείτε, Γάλλος βουλευτής αυτού του κοινοβουλίου τολμά να πει ότι το πρόβλημα το οποίο συνέβη στην Νορβηγία δεν ήταν σφαγή, αλλά ήταν η αφέλεια της νορβηγικής κυβέρνησης που δέχεται την πολυπολιτισμική κοινωνία, τότε πρέπει αυτό το κοινοβούλιο να πει ο κύριος Λεπέν είναι μια ντροπή για αυτό το κοινοβούλιο επειδή είπε αυτά τα λόγια. Et je voudrais Θα ήθελα να πω σε όλους τους πραγματικούς Ευρωπαίους Εάν αφήσουμε στα λόγια μας να περνάν αυτές οι φράσεις, εάν αφήνουμε να ακούγεται αυτή η ιδέα ότι η σημερινή Ευρώπη δεν μπορεί και δεν θα είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία, τότε όλοι μαζί ακολουθούμε τη γραμμή αυτών που κάνουν αποτρόπιες πράξεις. Υπάρχει πνευματική, διανοητική ευθύνη όλων μας όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Διότι δημιουργούμε το κλίμα, όπως είπε ο κ. Φερχόφστατ, δημιουργούμε ένα τέτοιο κλίμα όπου παράφρονες, τρελοί ενεργούμε αυτόν τον τρόπο. Το να σκεφτόμαστε την Νορβηγία σημαίνει να σκεφτόμαστε τι κάνουμε οι μεν και οι δε και τι λέμε οι μεν και η δε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς ε, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για διαφορετικά ζητήματα σε αυτή την ε, αίθουσα, αλλά νομίζω όλοι συμφωνούμε στο εξής. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος ανοχής, ελευθερίας και πλουραλισμού. Στο παρελθόν έχουμε πολεμήσει όσους δεν δέχονται την ανεκτικότητα, όσους ασκούν ε, καταπίεση και είναι κατά της δημοκρατικής μας κοινωνίας. Και τώρα και πάλι είμαστε κατά της εξάπλωσης του μίσους, του φόβου, της βίας. Δεν έχουν καμία θέση τα φαινόμενα αυτά στην Ευρώπη. Να εκφράσω εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας μου την βαθιά μου θλίψη για την απέσια αυτή βίαιη δολοφονία της 22 Ιουλίου. Πρώτα απ' όλα για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και για ολόκληρο τον νορβηγικό λαό και εξίσου σημαντικό για τους ε, σοσιαλιστές συναδέλφους στους οποίους ανήκαν οι νέοι που δολοφονήθηκαν, στην οικογένεια των οποίων ανήκαν οι νέοι που δολοφονήθηκαν. Εσείς ο ίδιος μας θυμήσατε, Πρόεδρε, την επέτειο της 9 ε, Σεπτεμβρίου, της ε, Σεπτεμβρίου πριν από λίγο. Να θυμίσω ότι πολύ καλά ακούστηκε και με ισχυρό λόγο ότι αυτοί οι τρομοκράτες διέπραξαν βίες πράξεις στο όνομα της θρησκείας αλλά εδώ είχαμε κάποιον που δεν εκπροσωπούσε καμία θρησκεία ούτε τους οπαδούς της. Η νορβηγική λοιπόν τραγωδία είναι κάτι ανάλογο το άτομο που διέπραξε αυτές τις δολοφονίες δεν εκπροσωπούσε κανέναν στην πραγματικότητα. Καμία θρησκεία, κανένα πολιτικό ρεύμα, απλώς το δικό του αρρωστημένο νου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προβάλλουμε, μάλλον να αντισταθούμε στον πειρασμό, να εκμεταλλευτούμε μια τέτοια ευκαιρία και να μην κάνουμε πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες επειδή αντιστάθηκαν πραγματικά στον πειρασμό αυτό. Η στάση τους ήταν αξιοπρεπής. Απέδειξαν ότι υπάρχουν ε, κοινέ αξίες που όλοι μοιραζόμαστε και τις οποίες μπορούμε να περασπιστούμε μαζί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Er Ευχαριστώ πολύ για την Νορβηγία. Μετά από τις 22 Ιουλίου ένα πράγμα είναι πλέον σαφές. Για μας ε, στην Σκανδιναβία αυτή η ημερομηνία σε πολλές πετυχέ ε, είναι η 11η Σεπτεμβρίου δεν ήταν τυχαίες αυτές οι πράξεις. Στόχευαν ακριβώς άμεσα την ίδια την Νορβηγία και την ίδια την δημοκρατία, το δημοκρατικό καθεστώς της Νορβηγίας, αλλά και κάτι παραπάνω ακόμα. Η επίθεση αυτή στην Όταγια είχε σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια ώστε να αποκεφαλιστεί η μελλοντική ηγεσία της σοσιαλδημοκρατίας στην Νορβηγία. Ήταν μια πράξη τρομοκρατική κατά του μέλλοντος. Η νεολαίοι αυτή του ε, σοσιαλδημοκρατικού κόμματος ε, ε, και ο στόχος αυτός δεν ήταν κάτι το τυχαίο. Αγωνιζόντουσαν κατά του ρατσισμού, υπέρ της ανεκτικότητας, υπέρ της ισότητας, υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, κατά της καταπίεσης, υπέρ της διεθνούς αλληλεγγύης ε, που ήθελαν να εκφράζουν οι πράξεις τους. Όλοι αυτοί οι νεολαίοι λοιπόν εκπροσωπούσαν ακριβώς εκείνο το οποίο περιφρονούσε με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο αυτός ο εγκληματίας τρομοκράτης. Η τρομοκρατική αυτή πράξη στον στιγερό της χαρακτήρα, στην φρικαλαιότητά της, δεν μπορεί να μας μάθει τίποτα, αλλά μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν ο ίδιος ο Πρωθυπουργό της Νορβηγίας και ο ίδιος ο λαός της Νορβηγίας. Άλλοι σε παρόμοιες ε, περιστάσεις θα ζητούσαν να υπάρξει εκδίκηση και θα είχαν διακηρύξει ένα πόλεμο κατά της τρομοκρατίας ε, περικόπτοντας τα δημοκρατικά δικαιώματα ε, άμεσα και οδηγώντας σε καταστολή. Και όμως δεν έγινε αυτό από πλευράς του Νορβηγού Πρωθυπουργού. Επέμεινε στο ότι η απάντηση σε αυτή την τρομοκρατική πράξη θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη δημοκρατία. Μεγαλύτερο δημοκρατικό άνοιγμα της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανθρωπιά και συμπόνια από την κοινωνία. Αυτή η στάση λοιπόν άξιζε την υποστήριξη και υποστηρίχθηκε από τον λαό της Νορβηγίας στο σύνολο της Νορβηγίας, στην Νορβηγία αλλά και στις άλλες ε, σκανδιναβικές χώρες αυτό το καλοκαίρι συναντήθηκαν εκατοντάδες ε, χιλιάδες, μυριάδες άτομα για να διαδηλώσουν κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας. Το μήνυμα όλων αυτών των διαδηλώσεων και των εκδηλώσεων ήταν σαφές ε, και αδιαμφισβήτητο. Το κακό μπορεί να σκοτώσει ένα άτομο, ποτέ όμως δεν μπορεί να νικήσει και να σκοτώσει έναν ολόκληρο λαό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε. παρακαλώ. Η ομάδα μου εκφράζει τη θλίψη της και την αλληλεγγύη της για την απόπειρα αυτή τη δολοφονική κατά του λαού της Νορβηγίας και κατά της ανθρωπότητας ολόκληρης. Πρόκειται για μια πράξη τελείως αδικαιολόγητη. Καμία ιδεολογία, καμία αιτιολόγηση δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς για να δικαιολογήσει μια σφαγή. Οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας και σε αυτό το αποτρόπαιο επεισόδιο θα πρέπει να βρίσκονται στο νου μας δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από τις αρχές στις οποίες βασίζεται η συνύπαρξή μας. Οι σχέσεις μεταξύ των λαών οι ίδιες. Ευχαριστούμε. Madame Diana Thank you, Mr. President. Um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όλοι μοιραζόμαστε τη λύπη, ε, το θυμό και την απελπισία μετά από αυτή τη μαζική σφαγή και θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου καθώς και των ψηφοφόρων μου για τον, ε, στο λαό της Νορβηγίας. Γνωρίζουμε στην περιοχή μου ποιος είναι ο τρόμος της τρομοκρατίας, αλλά δεν πρέπει ποτέ να στρέφεται προς τους νέους. Αυτό είναι ακόμα πιο αποτρόπιο και τρομακτικά. Πολύ, πολύ ε, μεγάλη ε, ε πολιτική, και άλλοι τοποθετήθηκαν. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ένα νέο ή μάλλον μία νέα που εξήγησε στο διαδίκτυο τι είχε κάνει. Έτρεξε, έτρεξε για να κρυφτεί και λέει «Ε, δεν, δεν καταλαβαίνω πώς σώθηκα ε, είμαι συντετριμένη και αναρωτιέμαι πώς επιβίωσα. Δεν μας άξιζε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τον νορβηγικό λαό. Νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Θα πρέπει ως δημοκράτες να δημιουργήσουμε ένα τείχο κατά της τρομοκρατίας και της βίας που δεν πρέπει να ε, αξιώνεται ποτέ ε, στην Ήπειρό μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συνέβη στις 22 Ιουλίου στην Ορβηγία είναι μια τραγωδία, μια βίαιη πράξη που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ούτε στα χειρότερα ε, στους εφιάλτες τους. Αυτός ο εφιάλτης όμως έγινε πραγματικότητα. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ε, στο... 80 άτομα έχασαν τη... Το άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το κρατικό κτίριο. Αργότερα όμως σκοτώθηκαν 70 νέοι. Αυτός είχε ε, δυθεί ως αστυνομικός. Και η αστυνομία, ο αστυνομικός είναι το σύμβολο της προστασίας και της ασφάλειας. Βεβαίω οι σκέψει μα βρίσκονται κοντά στην οικογένεια ε, των θυμάτων και στου φίλου του, αλλά και στον νορβηγικό λαό αλλά μας απασχολεί όλους αυτή η επίθεση, αυτή η σφαγή. Ήταν μια επίθεση κατά της δημοκρατίας, των δημοκρατικών θεσμών, των αξιών και των ιδεών μας. Ήταν μια επίθεση κατά νέων, οι οποίοι επρόκειτο να λάβουν ενεργό μέρος ε, στο δημόσιο βίο και στην πολιτική. Αυτά δείχνουν τον κίνδυνο των εξτρεμιστών. Επειδή αυτές οι ιδέες ενός παράφρονας άρρωστου καλλιεργούνται μέσω της ξενοφοβίας, του εξτρεμισμού, το, της επίθεσης κατά ε, μιας πολυπολιτιστικής κοινωνίας. Αυτή η ιδεολογία του μίσους είναι κάτι που πρέπει να καταδικάσουμε. Ο Νορβηγικό λαός με μεγάλη αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα αντιμετώπισε αυτά τα γεγονότα. Όλοι εντυπωσιαστήκαμε από τη δέσμευση του νορβηγικού λαού να σταθεί υπέρ τη δημοκρατίας, της διαφάνειας ε, ε, και των κοινών αξιών. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ας στηρίσουμε ενός λεπτού σιγή. Uh, Ήμην ε, των θυμάτων αυτής της φαγής. Της φαγής του Ιουλίου στην Ορβηγία. Πάμε πάλι στις πληροφορίες για να τις ολοκληρώσουμε. Ο συνάδελφος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να διαπιστώσω απλώς ότι ο κύριος Φάραλτ που βρίσκεται σε αυτό το κτίριο απουσίασε αντί να συμμετάσχει στο πένθος όλων των δημοκρατών που βρίσκονται στην αίθουσα της Ολομελίας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ατμόσφαιρα πένθους και θλίψης θα σας ενιστούσα να αποφύγετε να κάνετε προσωπικό.